της Ουκρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Προηγουμένως όμως, η κυρία Λίσα Φερέιρα παρετήθηκε. Κοινοποιούμε ότι η θέση έχει κενωθεί και ενημερώνουμε σχετικά τις εθνικές αρχές. Δεν έχω τροπολογίες όσον αφορά τις προτάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, όσον αφορά τις προτάσεις